Buenas tardes. Parece reanudamos la sesión. Αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας, είμαστε στο σημείο 8 της μεσημερινής διάταξης, ανταλλαγή απόψεων για το πολιτές σχέδιο για το απόθεμα το δικό απόθυμα σαφριδιού με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται σήμερα εδώ και θα κάνω μία σύντομη αναφορά σε αυτό το σχέδιο από το 2009. Έχουμε το σχέδιο αυτό και ε, είχαμε το 2009 μια προσανατολιστική ψηφορία, αλλά υπήρξαν κατόπιν αλλαγές και πραγματικότητα είναι ότι η Επιτροπή ψήφισε στις 26 Οκτωβρίου 2010 επίσημα και είχαμε και στις 23 Νοεμβρίου 2010 την ψήφιση της ε, έκθεσης, αλλά ελήφθησαν κάποιες πρωτοβουλίες ε, προκειμένου να γίνει επιπλοκή και ε, είχαμε και πρόταση συμβιβασμού από την Πολωνική Προεδρία ε, και το Φεβρουάριο του 2012 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από δύο προφορικές ρωτήσεις προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο και έναν τριμερή διάλογο άτυπο στις 8 Μαρτίου 2012. Σήμερα θέλουμε να ε, προωθήσουμε την έκθεση αυτή με την ακρόαση των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν διάφορες ιδέες. Καταρχήν θα σας ε, παρουσιάσω το πώς ε, θα οργανωθούμε. Έχουμε μία ώρα για τη συζήτηση. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλαχερ είναι εισηγητή για το πολιετέ ε, σχέδιο για το δυτικό απόθεμα του Σαφριδιού και κατόπιν ε, θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Προεδρία του Συμβουλίου και κατόπιν ε, στον εκπρόσωπο της ΓΑΜΑ ΜΑΡΕ και στη συνέχεια για 10 λεπτά θα πάρουν το λόγο οι δύο προσκεκλημένοι μας ο κύριος Αντωνίκη που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Πελαγικού ΡΑΚ και ο κύριος Μίλλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για ε, τους Εβραίους ε, διαδομένους πληθυσμούς ε, του Συμβουλίου για τη Διερεύνηση της Θάλασσας ε, και κατόπιν θα έχουμε μια συζήτηση με τους βουλευτές προκειμένου να θέσουν τις ερωτήσεις που επιθυμούν στους προκυκλισμένους και φυσικά θα μπορέσει να πάρει το λόγο και η Προεδρία τη Επιτροπή. Κύριε Γκάλακερ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. The reason I didn't respond, President, because... Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα θα ακούσουμε τους επιρρογνώμονες. Ε, και σίγουρα δεν είμαι εγώ. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, προτιμώ να μιλήσω τότε, αλλά χαίρομαι που η Επιτροπή δέχτηκε να οργανώσουμε αυτή την μήνυα ακρόαση και να προσκαλέσουμε τους ε, διακεκριμένους αυτούς ε, εμπειρογνώμονες. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι το Πελαγικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια κατήρθησε και δημοσίευσε την νομοθετική πρόταση ε, επί της οποίας ε, συντάσσω εγώ την έκθεση. Ήμουν εισηγητής το 2008 για πολλούς λόγους τροποποίησα την έκθεση μεταξύ των οποίων ε, διότι άλλαξαν οι κανόνες για τη συναπόφαση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, και δεν χρειάζεται τώρα να σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται με το Harvest Control Rule για οποιοδήποτε θέμα. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Από την άλλη πλευρά, πέρσι το Δεκέμβριο η πρόταση που κάναμε εμεί χρησιμοποιήθηκε ω τύπο για να προσδιοριστεί το ΤΑΚ σε, στην περιοχή ε, αυτή. Νομίζω καλύτερα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες ε, και στη συνέχεια μπορεί να υποφεληθώ τη ευκαιρία για να θέσω κι εγώ ερωτήματα. Πολύ ωραία. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο τη Προεδρία του Συμβουλίου, στον εκπρόσωπο τη Προεδρία του Συμβουλίου, αν θέλει τώρα να παρέμβει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, μιλήσω λίγο περισσότερο από τον ε, διακεκριμένο συνάδελφο Γκαλάχερ γιατί ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα για τη θέση μας. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ στην Επιτροπή και παρουσία εμπειρογνωμόνων έχουμε ήδη εκθέσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, από πλευρά της Δανικής Προεδρίας ε, με τιμά ιδιαίτερα που εκπροσωπώ εδώ το Συμβούλιο και έχω την ευκαιρία να σας εξηγήσω την θέση του Συμβουλίου για το Σαφρίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Κοινοβούλιο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, ούτω ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψει, να εξηγήσουν τι θέσει του και όπω είπε ο κ. Γκάλαχερ, ε, προσμένουμε στην Μήνυ ακρόαση για να ακούσουμε τους εμπειρογνώμενες από το Πελαγικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν ε, αρχίζοντας ε, να σας πω ότι σαφέστατα από πλευράς Δανικής Προεδρίας ε, θεωρούμε ότι είναι πρόσφορος ο διάλογος και κρίνουμε ότι θα είναι και επικοδομητικός ε, γιατί έχει σημειωθεί κάποια πρόεδρος ήδη από τον Μάρτιο. Το Κοινοβούλιο δέχθηκε επί της αρχής ε, κάποιες προτάσεις μας για τα θέματα ελέγχου. Τώρα είναι η περίοδος προβληματισμού για να περάσουμε στα δυσχερέστερα ζητήματα που σχετίζονται με το MSY, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το Harvest Control Rule, τον έλεγχο, το, τον έλεγχο των αλλιευμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσα στην αρχή. Πρόκειται για ε, την θέση της Επιτροπής αποκλειστικά και μόνο για το Σαφρίδη. Στη συνέχεια από το Πελαγικό ΡΑΚ και από την ISIS. θα ακούσετε ότι είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το ψάρι και άρα ε, ε, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και η θέση μας σε σχέση με αυτό το ψάρι. Δεν πρόκειται όμως για τα προγράμματα διαχείρισης, ούτε σχετίζεται η θέση θέση μας με την μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο διαφοροποίησε τη θέση του σε σχέση με την γενικότερη που ε, παρουσιάζεται την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποια επιμέρους στοιχεία ε, σε σχέση με το Σαφρίδι, τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Το πρώτο είναι ότι το άρθρο 43.2 θα είναι η νομική βάση και όχι το 43.3. Ε, στη συνέχεια, ο στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση βιώσιμης εκμετάλλευσης αυτού του αλλιεύματο επί τη βάση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ε, δυνάμει και των δεσμεύσεων πανέλου το 2002 Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιωάννεσμπουργκ. Στη συνέχεια, ε, μπορούμε να πούμε ότι ευθυγραμμίζεται με όλα τα σχέδια που εγκρίναμε από το 2007, παραδείγματο χάρη για τη Ρέγκα και το ε, Σαφρίδι, το, μάλλον το σχέδιο διαχείρισης του Σαφριδιού δεν διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα σχέδια και όταν προτείναμε αυτό το σχέδιο δεν υπήρχε το MSY μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, και στη συνέχεια προσαρμόσαμε το σχέδιο βάσει και αυτών που είχε εισηγηθεί η ISIS όταν καταθέσαμε την πρώτη πρόταση. Ε, λοιπόν, το σχέδιο όμως προβλέπει ευελιξία και βιωσιμότητα για το σχέδιο διαχείρισης βασιζόμενη στην εθνισιμότητα των ψαριών και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δηλαδή η εθνισιμότητα θα είναι κατώτερη του MSY με τρόπο ώστε να ε, υπάρξει σταθερότητα ε, στην διαχείριση του αλλιεύματος και από ό,τι κατάλαβα είναι από τις βασικές ανησυχίες του πελαγικού ΡΑΚ. Επίσης θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε το HCR, τον ε, έλεγχο των αλλιευμάτων μέσα στο σχέδιο. Θεωρούμε ότι για αυτό το απόθεμα που επί σειρά ετών ήταν κάτω του MSY δεν χρειάζεται εφαρμογή αυτού του κανόνα. Ε, περιοριζόμαστε λοιπόν στη μικροδιαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η προσέγγιση μα όμω δεν αποκλεί το HCR σε περιφερειακό επίπεδο βάσει τη αρχή περιφερειοποίηση. Αντίθετα, θα ευθυγραμμιζόταν απόλυτα με τα όσα έχουμε αποφασίσει για τα πολιετή σχέδια σχέδια διαχείρισης ε, που εγκρίναμε την περασμένη ε, εβδομάδα ε, ως προς τον γενικό κανονισμό στα πλαίσια της γενικής θέσης του Συμβουλίου σε συνεργασία με τους εταίρους μας όπως το πελαγικό ράκα προσυπογράψαμε και προτείναμε το HCR στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μόνη διαφορά είναι ότι το HCR δεν θα αποφασιστεί επί τη βάση συναπόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα χρειαστεί μικροδιαχείριση και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να αποφύγουμε τη μικροδιαχείριση σε επίπεδο Βρυξελών. Μπορώ να κατανοήσω την απογοήτευση του πελαγικού ΡΑΚ όταν διαπίστωσαν ότι διαγράψαμε το HCR, ενώ μετά από δυσχερέστερε διαπραγματεύσεις είχαν καταλήξει αυτό το αποτέλεσμα με τους εμπειρογνώμονες. Ε, δεν, δεν συμφωνούμε λοιπόν να αποφασίσετε αυτό επί τη βάση στην απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να συνοψίσω, και θα σταματήσω προς το παρόν για να μπορέσουν και άλλοι να τοποθετηθούν. Έχουμε λοιπόν σημειώσει πρόοδο για κάποια επιμέρους τμήματα του σχεδίου. Είμαστε ανοιχτοί για διάλογο, για τα εκρεμή ζητήματα και θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την περίοδο προβληματισμού με επικοδομητικό τρόπο, διότι ε, όλα όσα αποφασίζονται τώρα αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο Σαφρίδι και όχι σε άλλα πολυετή σχέδια ούτε για την ε, μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Δεν χρησιμοποιούμε το HCR βάσει του r 3 για το σχέδιο διαχείρισης του Σαφριδιού και η θέση μας για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση συνάδει με όλα τα υπόλοιπα σχέδια διαχείρισης που έχουμε εγκρίνει από το 2007 και μετά υπάρχει συνοχή. Δηλαδή θεωρούμε ότι το HCR επειδή βάζει την απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί σε μικροδιαχείριση. Γι' αυτό προτείνουμε την απαλληφή του κανόνα και χάρη στη θέση μας καλύπτουμε τις ανησυχίες περισταθερότητας ε, του πελαγικού ράκα και την ανάγκη να αλλιεύουμε κάτω από το MSY. Δεν αποκλείει η θέση μας ε, την ε, ε, θέσπιση HCR σε περιφερειακό επίπεδο βάσει της αρχής περιφερειοποίησης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσμένω στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το Πρόεδρε, όπως και οι υπόλοιποι ομιλητές, σας ευχαριστώ και εγώ για την οργάνωση της ακροάσεως που ελπίζω ότι θα επιτρέψει να διευκρινιστούν τα θέματα. Αν μου ζητήσετε να πω λίγα λόγια, εγώ θα περιοριστώ μοναχά σε δύο θέματα. Πρώτο, να πω ότι πράγματι, όπως εξήγησε ο εισηγητής, πρόκειται για πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην βάση των εισρωών των ενδιαφερομένων, του τομέα δηλαδή. Μετά από διαβούλευση και συνεργασία με αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο. Ο στόχος αυτών των ε, σχεδίων μακρόπνοης διαχείρισης είναι να εξασφαλιστεί η σταθερότητα για την υπεύθυνη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων προς το συμφέρον των ψαράδων, να έχουν δηλαδή τη βεβαιότητα για το μέλλον, μια προοπτική για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό δεν επιτρέπεται να το χάσουμε από τα μάτια μας ως στόχο. Κατανοώ τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους ενδιαφερομένους λόγω του χρόνου που παρήλθε μέχρι να καταλήξουμε στην παρούσα μορφή του φακέλου. Δεύτερο, η Κομισιόν από το 2009 προσπάθησε σε δύο περιπτώσεις να παίξει ρόλο του διαμεσολαβητή για να βρεθεί ένας συμβασμός. Και θα συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο αυτό κάθε φορά που μπορεί να βοηθήσει είτε από πλευρά Ένωση είτε από πλευρά Συμβουλίου. Και το 2011 άλλωστε και στην τελευταία Προεδρία η οποία κατέθεσε ένα πρώτο σχέδιο συμβιβασμού να είστε βέβαιοι ότι θα παίξουμε κατά το δυνατόν επικοδομητικό ρόλο. Για σήμερα προτιμώ να ακούσω τους εμπειρογνώμονες και το τι έχουν να πούν. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τους σημερινούς προσκεκλημένους. Καταρχήν να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Σένοντόνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν να αρχίσω, να πω ότι έχω ορισμένε διαφάνειες που απηχούν την ε, ομόφωνη θέση του πελαγικού ρακ και όχι μόνο του κλάδου, δηλαδή της βιομηχανίας, αλλά και οι μη κρατικές οργανώσεις μας υποστηρίζουν. Αυτά που θα παρουσιάσω σήμερα όπως είπα, είναι απήχηση ομόφωνης στάσης. Θα, δεν θα περιοριστώ μόνο στις καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν ήδη και που όντως μας έχουν απογοητεύσει και που θεωρούμε ότι το σχέδιο διαχείρισης που έχει υποβάλει το πελαγικό ΡΑΚ θα πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα περισσότερο αυτό και λιγότερο το MSY. Θα δούμε σε έναν αριθμό διαφανειών πολύ καθαρά γιατί καταλήγουμε στα συμπεράσματα που καταλήξαμε το 2009 και είχα ήδη κάνει τότε μια παρουσίαση στην Επιτροπή Αλίας σχετικά με το θέμα αυτό και οφείλω να πω ότι λάβαμε μεγάλη υποστήριξη από την Επιτροπή Αλίας για τα όσα κάναμε τότε. Πριν λοιπόν προχωρήσω στους βασικούς λόγους για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης, νομίζω είναι χρήσιμο για όλες και όλους να σας κάνω ένα ενσταντανέ ας πούμε σχετικά με το τι απασχολεί την αλία, τι σημαίνει οικονομικά και λίγες διαφάνειες σχετικά με το ιστορικό του σχεδίου διαχειρίσεως και πώς καταλήξαμε στην σημερινή ε, θέση του πελαγικού ΡΑΚ. Εδώ ομολογώ ότι ο συνάδελφος που θα με ακολουθήσει, David Miller, του έκλεψα μια διαφάνεια ε, και τον ευχαριστώ πολύ ε, για την διαφάνεια αυτή. Δείχνει εδώ ε, οι ροζ περιοχές είναι αυτές για τις οποίες μιλούμε, όπου είναι δηλαδή πολύ ε, ανεπτυγμένο το ψάρι εκεί. Θα δείτε και μια μικρότερη περιοχή με μοβ χρώμα. Αυτό είναι διότι όταν έγιναν οι εκτιμήσεις, ένα μέρος του αποθέματος μπαίνει στην ροζ περιοχή. Πάντως πρόκειται για ένα ελιστικό απόθεμα, απόθεμα το οποίο είναι πολύ εκτεταμένο. Δεν θα σας πω πολλά τεχνικά πράγματα, αλλά ένα πολύ σημαντικό θέμα για το σαφρίδι και ο λόγος δηλαδή που καταθέσαμε το σχέδιο διαχείρισης είναι ότι το ψάρι αυτό δεν ε, δεν βάζει τα αυγά του σε συγκεκριμένες πάντα περιοχές και σε συγκεκριμένο πάντα χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει κανείς. Το άλλο πράγμα που έγινε από τότε που φτιάξαμε το σχέδιο είναι ότι τώρα έχουμε σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπινη κατανάλωση του σαφριδιού. Προ 10 ετών δεν ήταν έτσι, δεν ήταν ανθρώπινη κατανάλωση. είναι σημαντικό, ε, σημαντικός τομέας οικονομικά. Να λίγα νούμερα σχετικά. Τα τελευταία χρόνια και χάρη στο σχέδιο φτάνουμε στις 180.000 τόνους περίπου αλίευμα με αξία σε πρώτη πόλη σε 125 εκατομμύρια ευρώ. Σε πράσινο χρώμα έχω βάλει ότι πριν από το σχέδιο διαχείρισης, 2009 δηλαδή, με νούμερα του 2007, η αξία πρώτης πώληση ήταν της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ, η δε τόνη που αλήβαμε ήταν 120.000. Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι έχουμε και έξτρα αλίευμα 60.000 τόνων, παρόλα αυτά καταφέραμε και διπλασιάσαμε την αξία του αλίευματος. Βασικός λόγος είναι διότι είχαμε σταθερότητα χάρη στο σχέδιο διαχείρισης. Υπάρχει μεγάλος, σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα πελαγικά σκάφη αλίας, είναι και μικρά σκάφη, βιοτεχνικά ας πούμε, και συνολικά πάνω από 600 σκάφη, 637 που ε, ανακατεύονται στην αλία αυτή. Ένα σύντομο ιστορικό του σχεδίου διαχείρισης Πριν από το, μάλλον μετά το 2003 δεν είχαμε αναλυτική επιστημονική παροχή συμβουλών. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις του Συμβουλίου και πάντοτε γινόταν συζήτηση για το πού θα βάλουμε τα ανώτατα ε, επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Δεν υπήρχε ωστόσο σταθερότητα για την πελαγική αλλία και δεν υπήρχε μακροπρόθεσμο, μακροχρόνιο σχέδιο. Το πελαγικό ΡΑΚ λοιπόν, λοιπόν, ήταν το πρώτο που είπε ότι χρειάζεται να πετύχουμε και την βιωσιμότητα και τη σταθερότητα. Υιοθετήσαμε λοιπόν τον Ιούλιο του 2007 το σχέδιο διαχείρισης βασισμένη σε μια πολύ καινοτόμα μέθοδο αξιολόγησης. Εδώ θα πω βέβαια σε τεχνικές λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι το σχέδιο βασίζεται σε ένα σταθερό συντελεστή 75.000 τόνων. Αυτά βασισμένα στο μέσο όρο τριών χρόνων και στην, ε, στις καταμετρήσεις αυγών σε βάθος ε, τριών ετών, όπως είπα. Αυτό μας δίνει βιωσιμότητα του αλλιεύματος, αλλά και ιδιαίτερα σταθερότητα στον κλάδο. Εμείς, όπως είπα, εγκρίναμε το σχέδιο αυτό τον Ιούλιο του 2007. Η ISIS το δέχτηκε ως προκαταρκτικό τον Νοέμβριο του 2007. Είναι ενδιαφέρον ότι τα ανώτατα επιτρεπόμενα αλλιεύματα από το 2008 έως το 2012 βασίζονται στο σχέδιο διαχείρισης και αυτό έχει δώσει μεγάλη σταθερότητα στην ε, αλλιευτική μας βιομηχανία. Να το λάβετε υπόψη σας αυτό όταν θα αποφασίσετε προς τα που θα, θα κατευθυνθείτε, δηλαδή θα βασιστείτε στο σχέδιο διαχείρισης ή στο MSY στο μέγιστο ε, βιώσιμο, ε, στη μέση, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και εκεί χρειάζεται βέβαια συμφωνία, το μάλλον η συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τώρα γιατί υποστηρίζουμε εμεί το σχέδιο διαχείριση. Για έναν αριθμό πολύ κέριων λόγων, ας πούμε η στρατηγική του διπλού S στα αγγλικά, δηλαδή βιωσιμότητα, sustainability του αλλιεύματος, διότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα το σχέδιο διαχείρισης αναπτύχθηκε με τη γνώμη των επιστημονικών συμβούλων και η ΆΙΣΕΣ το δέχθηκε προκαταρκτικά, διότι ε, εξασφαλίζει την βιωσιμότητα. Ο δεύτερος κέριος παράγοντας είναι ότι προσφέρει σταθερότητα στην αλληλευτική βιομηχανία και αυτό εννοώ όταν λέω διπλό S, δηλαδή sustainability και stability στα αγγλικά. Βέβαια μια εικόνα αξίζει χίλια λόγια αυτό που θα ήθελα να συγκρατήσετε από την ε, παρουσίασή μου είναι αυτός ο πίνακας. Εδώ θα σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα, κοιτάξτε τις γαλάζιες κάθετες γραμμές που απηχούν τις επιστημονικές συμβουλές της ISIS πριν από την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ευφυΐα για να καταλάβει ότι το πράγμα πήγαινε πάνω κάτω. Μια πάνω, μια κάτω. Εδώ το δεύτερο που έχω βάλει είναι τα χρόνια όπου άρχισε να χρησιμοποιείται το σχέδιο διαχείρισης για τα τάκ και τις ποσοστώσεις και εκεί έχει αλλάξει πολύ λίγο η απόδοση και αυτό εννοώ όταν, λέω για βιωσιμότητα, όταν μιλώ για βιωσιμότητα και για σταθερότητα και το τελευταίο που θέλω να σας τονίσω είναι αποφασίσαμε αν είχαμε αποφασίσει μάλλον να δεχτούμε την στρατηγική της, ε, του, του, της μέγιστης βιωσιμο, βιώσιμης απόδοσης που ζήτησε το Συμβουλίο, θα είχαμε αυξήσει κατά 21% τις καταβολές και φέτος, τον προηγούμενο χρόνο και φέτος 13%. Και θα με ρωτήσετε γιατί, θα εκπλαγείτε γιατί ο κλάδος δεν δέχτηκε τις αυξήσεις αυτές δεν ζεχτήκαμε, διότι συμφωνήσαμε όλοι ότι με το σχέδιο διαχείρισης εξασφαλίζαμε την βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του κλάδου. Έτσι, εάν εξετάσετε το αριστερό τμήμα, αλλά και τις πράσινες γραμμές του MSY, θα δείτε ότι κάθε χρόνο πάλι θα ανεβοκατεβαίνουμε και θα καταστρέψουμε τη σταθερότητα που έχουμε εξασφαλίσει για την ε, αλληλευτική βιομηχανία. Το γράφημα σας δείχνει καθαρά για ποιο λόγο εμείς ως πελαγικό ρακ ομόφωνα θέλουμε να διατηρήσουμε τους κανόνες του σχεδίου διαχείρισης. Το άλλο που πρέπει να σημειώσετε είναι ότι ακολουθούμε την δήλωση πολιτικής της Κομισιόν πρόσφατη που λέει ότι θα πρέπει να ακολουθούν τα σχέδια διαχείρισης όπου υπάρχουν τέτοια. Και αυτό είναι το βρίσκω πολύ σωστό. Δεύτερο, ότι το σχέδιο διαχείρισης υποστηρίζεται από την ίδια την τεχνική, επιστημονική και οικονομική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμορφώνεται με το πλαίσιο της ε, μέγιστης βιώσιμης ε, απόδοσης, γίνεται δεκτό ως προκατακτικό μέτρο από την ISS, βραχυπρόθεσμα δηλαδή τουλάχιστον, και είμαι σίγουρος όταν, όταν ο συνάδελφος της ISS θα σας πει ε, τα δικά του, θα σας πει κιόλας ότι και η ISS ετοιμάζεται να κάνει προτάσεις για μακρόχρονη σταθερότητα. Θα ολοκληρώσω με δύο παρατηρήσεις. Το πελαγικό ΡΑΚ βρίσκεται στην πρωτοπορία για να διορθώσει ένα σύστημα το οποίο δεν, δεν λειτουργούσε. Θυμηθείτε το γράφημα που σας εξήγησα με τις χρωματιστές γραμμές που προτείνει ένα βιώσιμο μακροπρόθεσμο ε, πρόγραμμα διαχείρισης, σχέδιο διαχείρισης για το Σαφρίδι. Γιατί άραγε να προσπαθήσουμε, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, να χαλάσουμε ξανά το σύστημα εγκρίνοντας, υιοθετώντα μια διαφορετική προσέγγιση στην βάση των MSY των ε, μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων. Ελπίζω να δεχτείτε την άποψη του πελαγικού ΡΑΚ. Ίσως να σας φαίνεται βολικό να λύσετε το πρόβλημα του άρθρου 42.2 και 43.3, δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά σίγουρα αυτό δεν λύνει το πρόβλημα από την άποψη του πελαγικού ΡΑΚ. Ε, ζητώ συγγνώμη, μακρηγόρησα κάπως, αλλά αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μίλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Λέγομαι David Miller, ε, είμαι ερευνητή ε, στο ε, Ινστιτούτο για τι Μελέτε Οικοσυστημάτων στι κάτω χώρες και ε, είμαι πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας WGY. Είναι μια ομάδα εργασίας ε, αξιολόγησης που ασχολείται με τα εκτεταμένα και αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα. Και η δουλειά μας είναι να έχουμε δεδομένα για να αξιολογήσουμε τα επίπεδα της εκμετάλλευσης και να δίνουμε κάποιες συμβουλές ε, για την ε, αλία. Επίσης, ε, έχω δώσει συμβουλές για τα πελαγικά αποθέματα και για τη Βόρεια Θάλασσα και έχω, και έχω αξιολογήσει κάποιες στρατηγικές διαχείρισης στον Καναδά και έχω εμπειρία με, με σχέδια διαχείρισης στην Νότια Αφρική, στο Cape Town. Σήμερα διαχειριζόμαστε την αλία βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Η ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι μια έννοια η οποία ουσιαστικά είναι σαν να ε, βρίσκεται ο χρυσός ε, στην άκρη του ουράνιου τόξου. Δηλαδή φαίνεται να είναι μια ωραία ιδέα, αλλά για μια, πρακτικούς λόγους, όπως και για κάποια αποθέματα, όπως το δυτικό απόθυμα του Σεφριδίου, είναι κάτι που ποτέ δεν θα πετύχουμε, συνεχώς το κυνηγάμε και προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε στη μέγιστη βιώσιμη αποδοσή. Και όταν όσοι έλαβαν τι αποφάσει το 2002 στο Ιωάννεσμπουργκ προσπαθήσαν να αποφασίσουν πώ θα γίνει τη διαχείριση τη αλεία, εξέτασαν την έννοια τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και είδαν την αξία που υπάρχει εκεί. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη βιώσιμη αλεία και για να έχουμε μια, ένα καλό κλάδο και θέλουμε να είναι βιώσιμο όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για ε, την ίδια την αλεία. Έτσι λοιπόν λοιπόν μέγιστη ε, απόδοση σημαίνει ότι το απόθεμα θα είναι σε τέτοια κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν μιλάμε για υπερεκμετάλλευση του αποθέματος αλλά θέλουμε να έχουμε υγεία αποθέματα και να μπορούμε να αλλιεύουμε στο δυνατόν περισσότερο από το απόθεμα αυτό. Στην ε, ε, πράξη μπήκε αυτή η έννοια στην νομοθεσία και προσπαθήσαμε να την εφαρμόσουμε με έναν πρακτικό τρόπο. Προσπαθήσαμε να ορίσουμε τι είναι μέγιστη βιώσιμη απόδοση και πώς θα φτάσουμε εκεί. Και σε ό,τι αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορείτε να δείτε τρία διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε το ίδιο το μεσουάι που είναι το αλλιευμά και το πιο επίπεδο αλλιεύματος ε, ε, που θέλουμε να φτάσουμε. Έχουμε το BMSY που είναι βιομάζα που σχετίζεται με αυτό το ελίευμα και αυτό σημαίνει σε ποια κατάσταση πρέπει να είναι το για να έχουμε υψηλό ελίευμα και είναι και το FMSY που είναι το ποσοστό της εκμετάλλευσης του αποθέματος και αυτό είναι διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα, εξαρτάται δηλαδή από το ποια είναι η κατάσταση του αποθέματος. Έτσι λοιπόν, ε, όταν ε, θέλουμε να καθορίσουμε την πολιτική για την εφαρμογή τη Συμβουλή για το MSY, αποφασίσαμε να έχουμε το FMSY, που είναι το ποσοστό εκμετάλλευση, το οποίο θα μα δώσει τη μέγιστη δυνατέ αποδόσει, ενώ δεν θα το απόθεμα και σε μια υγιή κατάσταση. Και αυτό έχει νόημα γιατί και το BMSY και το BMSY ε, είναι έννοιες ισορροπίας. Έτσι λοιπόν, μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να έχουμε ε, το μέσο όρο του ελλείμματος ή της βιομάζας ε, που προκύπτει. Σε ένα δεδομένο έτος, κυρίως σε βραχυπρόθεσμα, θα έχουμε περιβαλλοντικές αλλαγές, αλλαγές στη μετανάστευση του αποθέματος, στην τροπολία και μπορούν πολλοί να είναι οι παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στο ποια θα είναι η κατάσταση του αποθέματος σε ένα συγκεκριμένο έτος. Έτσι λοιπόν ε, θα υπάρχει μια λογική διακύμανση. Έτσι λοιπόν το FMSY είναι μια βιώσιμη προσέγγιση για να ακολουθήσουμε. Το πρόβλημα είναι σε ό,τι αφορά το δυτικό πόθεμα σαφριδίου ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Όταν ε, πριν ε, ε, από χρόνια είχαμε την ε, ε, βιομάζα των εμπορικών ποθέματος. Αυτό μας δείχνει το μέγεθος του ποθέματος και αριστερά έχουμε την ανασύσταση, δηλαδή τον νέο πληθυσμό που μπαίνει στο απόθεμα κάθε χρόνο. Και όπως βλέπετε σε αυτή την σχέση κάθε χρόνο δεν υπάρχει πολύ μεγάλο σχετισμό και για να έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη αποδόση θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του αποθέματος που θα μου δώσει υψηλή ανασύσταση. Αυτό καλούμε εμείς παραγωγικότητα στην αλία, δηλαδή ποιε νέε δραστηριότητες μπαίνουν στην αλήψη κάθε χρόνο. Και έτσι λέμε, αν έχουμε χαμηλό απόθεμα, ε, τότε θα έχουμε χαμηλή ανασύσταση. Όμως ε, εδώ έχουμε ε, πολύ χαμηλές βιομάζες και έχουμε τη μέγιστη δυνατή ανασύσταση και βλέπουμε ότι έχουμε χαμηλή ανασύσταση. Έτσι λοιπόν το να έχουμε ένα μεγάλο απόθεμα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη ανασύσταση και να έχουμε ένα μικρό απόθεμα, όσο μικρό το είδαμε, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και μεγάλη ανασύσταση. Δεν αποτελεί εγγύηση. Όμως ε, ε, ποτέ το απόθεμα δεν έφτασε πολύ κοντά στα όρια εμείς ε, μπορεί να φτάσουμε τελικά να έχουμε ε, την χαμηλή ανασύσταση και να έχουμε βλάβη της ε, παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν, τι λέμε, για να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το FMSY δεν την χάνει ικανοποιητική εκτίμηση για το σαφρίδι. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε το FMSY και το STCF, ε, ε, το ΕΑ έχει ήδη σημειώσει ότι αυτή η αρχή δεν είναι αρχή της πρόληψης. Σε ό,τι αφορά τώρα το πλαίσιο του ISIS, ε, πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το σημείο αναφοράς και έχει να κάνει με την αξιολόγηση του αποθέματος και για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού. Όπως φαίνεται είναι ευρέα διαδεδομένο και μετακινείται. Έχει πολλές περιοχές ανασύστασης προσπαθώντας ε, να έχουμε ένα δίκτυ για όλο το απόθεμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τι κάναμε. Κάθε τρία χρόνια πάμε στον ωκεανό και προσπαθούμε βάσει των αυγών να δούμε πόσα ψάρια υπάρχουν. Όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι και πολύ ακριβές, όμως παρόλα αυτά είναι ένας καινοτόμος τρόπος για να έχουμε κάποιες ενδείξεις σε σχέση με το ποιο είναι η κατάσταση του αποθέματος. Όμως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αυτές τις εκτιμήσεις μόνο κάθε τρία έτη. Είναι πολύ αραιά τα στοιχεία που έχουμε. Έχουμε αυτό τον ε, ε, ανεξάρτητο δίκτυ της αυθονίας μόνο κάθε τρία έτη. Έτσι λοιπόν τι συμβαίνει εδώ. Οδηγείται σε τήσεις αλλαγέ ε, στο επίπεδο του αποθέματος όπως έχει εκτιμηθεί. Όταν κάνουμε αξιολόγηση του αποθέματος δεν έχουμε δεδομένα από ένα έτη πόσα ψάρια υπάρχουν έτος και τελικά ολοκληρώνουμε την όλη διαδικασία. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ευρύτερο, δηλαδή να έχουμε κάποια δεδομένα. Παραδείγματο χάρη, είδαμε πόσα ψάρια είχαμε που ήταν 7 ετών το 2007, ε, πόσα ψάρια 5 ετών είχαμε παραδείγματο χάρη το 2006 κτλ. Έτσι ώστε έχουμε νέα δεδομένα κάθε έτος. Δεν αλλάζει την αντίληψή μα για το που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με πέρσι, Απλώ αλλάζει όλο το ιστορικό σε σχέση με το πώ αντιλαμβανόμαστε το απόθεμα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι είναι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι βάσει των πιο πρόσφατων δεδομένων και των πιο πρόσφατων πληροφοριών δεν μπορούμε να εγγυθούμε τι συνέβαινε πριν πέντε χρόνια, παρά μόνο να έχουμε περισσότερα δεδομένα που θα φτάσουν σε εμά. Ένα πρόσθετο πρόβλημα με την σε χρήση των αξιολογήσεων και την παροχή συμβουλών είναι ότι οι εκτιμήσει των πλέον πρόσφατων χρόνων των αξιολογήσεων, δηλαδή ε, ε, ε, είναι τα έτη που είναι τα πιο βέβαια, μας ρωτήσετε ποια ήταν η βιομάζα το 95, Μάλλον θα σας πούμε κάτι φέτος που θα μοιάζει με αυτό που θα σας πούμε του χρόνου και του παραχρόνου. Ενώ αν μας ρωτήσετε για τη βιομάζα το 2010, αυτό που θα σας πούμε φέτος θα μπορούσε να διαφέρει από αυτό που θα σας πούμε το 2013 και θα σας πούμε το 2014. Έτσι λοιπόν είναι αβέβαιες οι αξιολογήσεις μας δεν θα μπω σε λεπτομέρειε γιατί, αλλά επειδή έχουμε αιτήσει αλλαγέ στην αντίληψη του αποθέματο και ιδίω τα τελευταία έτη, σημαίνει ότι αν έχουμε συμβουλέ που βασίζονται σε αιτήσει αξιολογήσει, είναι πιθανό να έχουμε συμβουλέ που ποικίλουν, να διακυμαίνονται όχι μόνο επειδή αλλάζει το ίδιο το απόθεμα, αλλά επειδή αλλάζει και την μια αντίληψη για το απόθεμα. Έτσι λοιπόν είναι αρκετά δύσκολο να προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε τι κάνουν τα ψάρια όταν ε, υπάρχει και επιστημονική αβεβαιότητα και τη βάζουμε μέσα στις διακυμάνσεις του ελιεύματος. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό. Έχουμε λοιπόν ε, τους κανόνες ελέγχου του αποθέματος. Ε, θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες, δεν θα σας πω λεπτομέρειες για τις αξιολογίες που κάναμε. Δεν ε, θα το κάνω αυτό. Έχω προετοιμάσει μια άλλη παρουσίαση, πολύ πιο τεχνική και καλύπτει πάρα πολλέ από τι λεπτομέρειε που κάναμε τελευταία πεντέτη και αν θέλετε θα σα τη δώσω. Αλλά το 2007 κάναμε κάποιες αξιολογήσεις ε, όπου είδαμε τον HCR τον κανόνα αυτό της εκμετάλλευσης του αποθέματος και ακόμη και αν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε παρκώς ε, την αυθονία του 2006, αν δείτε όλο το ιστορικό της εξέλιξης του αποθέματος, έχετε μια καλύτερη ιδέα για την δυναμική του αποθέματος. Έτσι λοιπόν, δεν ε, είναι απαραίτητα η αυθονία που κοιτάμε, αλλά αξιολογούμε το σχέδιο της διαχείρισης και τον HCR ε, για να κατανοήσουμε τη δυναμική και μπορεί να υπάρχουν νέα δεδομένα που θα αλλάξουν την αντίληψή μας πολύ συχνά, υπάρχουν και κάποιες σταθερέ, Έτσι λοιπόν, λοιπόν όταν ε, δοκιμάζουμε τη στρατηγική διαχείριση μπορούμε να δούμε πώ αυτό έχει αντίκτυπο στο αλλίευμα, στην παραγωγικότητα και αν το δούμε με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχουμε διαχείριση μακροπρόθεσμα βάση, μακροπρόθεσμα βάση μακροπρόθεσμων στόχων αλλά μπορείτε να αξιολογήσετε την επίδοση του HCR έναντι των μακροπρόθεσμων στόχων. Και τι εννοώ είναι ότι η διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές τη ε, της τη βιώσιμη αποδοση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να χρησιμοποιούμε καπευθεία σημεία αναφορά μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το MSY κάθε χρόνο για να πετύχετε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Μπορείτε να το κάνετε με έναν ε, πιο έμεσο τρόπο και μακροπρόθεσμα να ελέγξετε αν σα δίνετε αποτελέσματα που θέλετε. Έτσι λοιπόν τελικά πρέπει να αποφασίσετε μεταξύ ενό κανόνα εκμεταλλεύση του καθποθέματο που έχει δοκιμαστεί ε, και, ενός, και μια μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, που δεν έχει καθοριστεί όπω πρέπει και εμεί θέλουμε να προτιμούμε τον HCR. Όταν κάνετε μια νέα αξιολόγηση, ε, αξιολογούμε ε, χρησιμοποιώντα και το πρόξι τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Βέβαια, αυτό ακόμη δεν το έχουμε πράξει. Έτσι λοιπόν, ένα σχέδιο διαχείριση μπορεί να βελτιστοποιήσει το ελιευμά και να ελεγχιστοποιήσει το κίνδυνο του αποθέματος, αλλά χωρίς ε, να χρησιμοποιούνται αυτοί οι δύο κανόνες το ίδιο το HCR. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι ε, μία στάνταρ πρακτική είναι ότι πρέπει να επεξιολογούνται τα πράγματα κάθε 3-5 έτη, καθώς ε, προκύπτουν νέα δεδομένα και νέα γνώση και αν είχε γίνει αποδεκτό αυτό το σχέδιο αμέσως, τώρα θα είχαμε φτάσει στην επανεξιολόγηση. Και όπως το βλέπω, είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε αυτό τώρα, έχουμε νέα πλατφόρμα αξιολόγηση για να το πράξουμε αυτό με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο ίσω. Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και του συναδέλφου που με βοήθησαν ε, με τη δουλειά αυτή από το Ηνωμένο και την Ιρλανδία και τι κάτω χώρε και όλη την ομάδα εργασία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μίλλερ. Να περάσουμε τώρα, να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές που θέλουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Κυρία Λοβέν, κάποιος άλλος θα πάρει το λόγο για να απολογίσουμε το χρόνο. Παρακαλώ ζητήστε τώρα το λόγο. Καταρχήν κυρία Λοβέν. Okay. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους δύο μιλητές γιατί ήταν διαφωτιστικότατοι ε, σχετικά με τη θέση του Πελαγικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ε, ήταν παιδαγωγική η μέθοδός σας και καταδείξατε ότι για τη βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύουν ε, σταθεροί όροι για το μέλλον και να μην πέφτουν θύματα της διακύμανσης ανάλογα με τις επιστημονικές συμβουλές και τις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ακριβώς το μήνυμα επιθυμώ να περάσω και εγώ και γνωρίζω το ίδιο ισχύει και για τον γάδο στην ε, Βαλτική. Αν εφαρμοστεί εκεί το, η προσέγγιση FMSY αποκλειστικά και μόνο θα είχαμε ε, συν 40% πέρσι, ενώ τώρα περιορίζεται αυτή η αύξηση από ε, το πολιετές σχέδιο, έχοντας έτσι ένα συν πλήν 15% και εξασφαλίζοντας σταθερότητα για τον κλάδο. Αυτό αποδεικνύεται λοιπόν από τους επιστήμονες ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά υπάρχουν ε, στοιχεία που δεν γνωρίζουμε, για τα οποία δεν είμαστε σίγουροι για, ως προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς το FMSY ετησίως. Δεν μπορούμε όμως ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό ως πρόσχημα για να μην συμμορφωνόμαστε με τις επιστημονικές συμβουλές. Θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ε, ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε την προληπτική προσέγγιση και να έχουμε επίπεδα αποθέματος Ευχαριστώ άνω αυτών που μπορούν να μας ε, προσφέρουν ε, το MSY τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Χαίρομαι λοιπόν που και οι επιστήμονες του ISIS μας ε, επιβεβαιώνουν ότι δεν μπορούμε να κοιτάζουμε, να εξετάζουμε ένα έτος μόνο για να καταλάβουμε ποιο είναι το MSY. Πρέπει να κοιτάξετε προς τα πίσω 3-4 χρόνια για να καταλάβετε τι αποτέλεσμα έχει χρήση του MSY και είναι καθήκον Λοιπόν των πολιτικών να εφαρμόζουν την προληπτική προσέγγιση διότι είναι η ευνοϊκότερη λύση, το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον κλάδο ούτω ώστε να έχουν και μελλοντικά σταθερότητα. Λοιπόν, ε, είμαι πραγματικά ευγνώμων προ ε, τον εισηγητή μα, ε, τον κύριο Γκάλεχερ, που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και προ του ομιλητέ, διότι αυτό δείχνει ακριβώ την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε κατά τη μεταρρύθμιση κοινή ελευτική πολιτική. Χρειαζόμαστε δηλαδή πολιετή σχέδια διαχείριση και την προληπτική προσέγγιση. Φτάνω στο δεύτερο σημείο. Η τωρινή κατάσταση ε, σε σχέση με το Συμβούλιο για τις κανόνες εκμετάλλευσης και όλα αυτά. Νομίζω ότι και οι δύο μιλητέ ε, πέραν κάθε αμφιβολία ξεκαθάρισαν ότι το να χρησιμοποιήσουμε μόνο και μόνο το FMSY στο πολιετέ ε, διαχειριστικό σχέδιο δεν επαρκεί διότι έτσι υπάρχει ε, κίνδυνος μεγάλων διακυμάνσεων της ε, θνησιμότητας ε, διορθώνει μιλήτρια των ουσιαστικών αλλιευμάτων και φυσικά είναι απευκταίο αυτό, άρα ναι, αυτό που θα ήθελα τώρα είναι να ακούσω την απάντηση του Συμβουλίου μετά από αυτές τις δύο παρουσιάσεις θεωρεί το Συμβούλιο ότι ε, είναι καλό να υπάρχουν τόσο μεγάλες ε, διακυμάνσεις ε, στα αλλιεύματα. Πώς προτείνει το Συμβούλιο, τι προτείνει το Συμβούλιο σε σχέση με την προληπτική προσέγγιση. Δεν έχω λοιπόν άλλε ερωτήσεις. Κλείνω συγχαίροντας και τον εισηγητή και τους δύο μιλητές. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Όχι, τότε Συμβούλιο Επιτροπή. κάποιο από του συγητέ, ε, από του προσκεκλημένου, όπως θέλει κάτι να διευκρινίσει. Señor Gallagher, me ha pedido la palabra. Κύριε Γκάλακερ, θέλετε το λόγο. Να προσθέσω και εγώ κάτι σε σχέση με αυτά που μόλις ακούσαμε. Κατεδείχθη και από τον κύριο Μίλε και τον κύριο Ντόνικ ότι είναι μονόδρομος αυτός ο κανόνας εκμετάλλευσης, το HCR. Έχω πει στο παρελθόν ότι για να έχουμε το HCR ε, θα πρέπει να αυξήσουμε κατά 15% τα τάκαλα στα αριθμητικά στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος και βλέπουμε ότι το 2011 αν είχαμε δεχτεί τότε ε, το HCR και όχι το MSY θα είχαμε συν 21% στο απόθεμα του Σαφριδιού. Το 2011 αν το είχαμε δεχτεί θα είχαμε άλλα 13%. Ε, Αυτό θέλουν ε, οι αλληλείς. Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αλληλείς, είναι και επιχειρηματίες και συνειδητοποιούν ότι το εισόδημά του ε, πρέπει να το εξασφαλίσουν μακρόπνοα γιατί συνεργάζονται με τι τράπεζε, Οι τράπεζε λοιπόν θέλουν να γνωρίζουν επίση τι σκοπεύουμε εμεί να κάνουμε με τα ε, πολιετή σχέδια διαχείρισης ε, και νομίζω ότι ο κύριο Τίμισον το έχει πει αυτό πολλέ φορέ στο παρελθόν. Θέλουν παραδείγματο χάρη να ανακοινήσουν το σκάφο ή να αγοράσουν νέο. για να ληφθούν τέτοιε αποφάσει χρειάζεται ένα πολιετέ σχέδιο διαχείριση. Άρα είναι προφανέ προφανές ε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε εφ' ε, και ήθελα να πω ότι τις τελευταίες ε, ημέρες είχαμε πολύ καλή συνεργασία με το Συμβούλιο αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε τους, μέσα από τους τριμερείς διαλόγους θα σημειώσουμε πρόοδο και είχαμε και έναν σε σχέση με την έκθεση αυτή νωρίτερα το 2012 κατεγράφει κάποια πρόοδο, όχι η επιθυμητή, αλλά Αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι θα λήξει η ιδανική προεδρία σύντομα. Γνωρίζετε πάντως ε, ότι Προτού τελειώσει ο μήνας θα μπορούσατε να αφήσετε ένα κληροδότημα για την Κυπριακή Προεδρία, η οποία σίγουρα θα έρθει να μας συναντήσει για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Δεν θέλω να είμαι κοινικός, αλλά ε, το θέμα είναι το 42-2 το 43-3. Εφόσον έχουμε αρμοδιότητα ε, συναπόφασης, ε, δεν θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μόνο το άρθρο. υπάρχουν ναι, και άλλες παράμετροι και ούτως ή άλλως στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε τα τάξη και οι ποσοστώσεις να προσδιορίζονται βάσει συναπόφασης. Εμείς θα ορίζουμε τις παραμέτρους βάσει των οποίων θα λαμβάνεται η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ελπίζω λοιπόν να διευκρινιστούν κάποια ε, σκοτεινά σημεία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλαχερ. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιο άλλο το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι τους δύο προσκεκλημένου μας σε αυτή την μήνυα κρόση και να συνεχίσουμε με τα εργασία τη Επιτροπή μας. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξη, Εξωτική διάσταση της κοινή ελευτική πολιτική. Η κυρία Λαβέν είναι η συγγήτρια. 8 Μαΐου ήταν η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Έχουν παρουσιαστεί 284 τροπολογίες. Είχαμε συζητήσει στις 21 Μαΐου τις τροπολογίες και σήμερα θα έχουμε τη δεύτερη συζήτηση Ιδίω για τις συμβιβαστικές τροπολογίε, γνωρίζοντας ότι η ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για τη συνεδρία τη 11η Ιουλίου. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοβέν. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου για τις τροπολογίες που κατέθεσαν, που όπως είπατε είναι πολλές. Μια στιγμή παρακαλώ διακόπτη πρόεδρος να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι άνθρωποι με ησυχία. Thank you. Go ahead. Thank you. Ωραία, συνεχίστε. Ναι, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ καλύτερα τώρα. Καλά, κοιτάξτε. Στο Στρασβούργο κάναμε μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών και των όσων είχαν καταθέσει τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη από τις και τους συναδέλφους, διότι όσο γνωρίζετε υπήρχε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τον βασικό κανονισμό που έλεγε τη Δευτέρα και μετά υπήρχαν και οι λίστες ψηφοφορίας για την αγορά που ψηφίσαμε σήμερα. Φαίνεται να μην έγινε πολύ πρόοδος από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και τότε προτάθηκαν συμβαστικές τροπολογίες. Υποτίθεται ότι θα είχαμε κάποιες απαντήσεις για τις τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες, αλλά δεν έγινε αυτό. Οι προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες εξακολουθούν να είναι οι ίδιες που ε, θα έχουμε περισσότερες συμβαστικές αυτή την εβδομάδα και ελπίζω να ξανασυναντηθώ με τους ε, σκιώδεις ηγητές τη μεθ' επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν οι βασικά οι συμβιβαστικέ τροπολογίες φαίνεται πως ε, υποστηρίζονται, θα τις περάσω σύντομα και μετά να μπορέσουν να συζητήσουν οι συνάδελφοι. Έχω δύο ξεχωριστές συμβατικές, μία για το recital ε και μία για την παράγραφο 4, όπου το ίδιο πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να μείνει μια αιτιολογική σκέψη που να μιλεί για πολιτική για την ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως ορισμένες τροπολογίες που μιλούν για συνοχή πολιτικής και σε πολλούς άλλους τομείς πολιτικής όπως εμπόριο, ε, περιβάλλον, ε, υγεία κλπ. Και στρατηγική Ευρώπης 2020 Νομίζω ότι είναι καλό να μείνει ως μία παράγραφος, γιατί πρόκειται για τη συνοχή της πολιτικής που περιλαμβάνεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας και μιλώ για το άρθρο 208 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους ε, συνεργασίας για τις ε, ε, πολιτικές εκείνες οι οποίες έχουν, σχέση με χώρες υπό ανάπτυξη. Και βέβαια εδώ το θέμα θίγει πολύ τι αναπτυσσόμενε χώρε. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλύτερα να μείνει η αιτιολογική σκέψη καθαρή, ξε, ε, σκέτη και να έχουμε μια άλλη αιτιολογική σκέψη που να μπουν μέσα όλες οι πολιτικές που πρέπει να συντονιστούν και που έχουν σχέση βέβαια με χώρε που δεν είναι μέλη τη Ένωση. Φαίνεται ότι αυτές υποστηρίζονται οι συμβαστικές τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, υπάρχει και μια συμβιβαστική που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με μεγάλη υποστήριξη από ό,τι φαίνεται. Και ένα κέριο θέμα της μετακίνησης από σημαία σε σημαία των σκαφών. Η παράγραφος πρότεινα εγώ έχει τροποποιηθεί από ορισμένου συναδέλφου. Έχει τροπολογηθεί καλύτερα. Και εμεί προτείνουμε, εφόσον ένα σκάφο φύγει από το νεολόγιο μια χώρα μέλου για να πάει να ψάξει να βρει αλληλευτικέ ευκαιρίε αλλού, να μην μπορεί να επωφελείται για 24 μήνες των πλεονεκτημάτων που έχουν τα σκάφη της ένωση λόγω των σχετικών συμφωνιών. Φαίνεται ότι γι' αυτό υπάρχει υποστήριξη. Έχουμε και άλλη συμβιβαστική για τα RFMO που βασίζονται ε, η αρχική παράγραφος έλεγε ότι θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα απλουστευτικά κριτήρια των ιστορικών αλλιευμάτων, αλλά κυρίως σε κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Και μιλώ για τις περιφερειακές, διαχειρήσεις, ε, περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας. Βέβαια, τα ιστορικά αλλιεύματα είναι ένα κριτήριο, αλλά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και βεβαίως και οι θεμητές προσδοκίες των χωρών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη όταν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλληλείας θα αναπτύσσουν τα συστήματά τους. Επίσης υπάρχει μία όπου θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Να αλλάξουμε δεύτερη δηλαδή την παράγραφό μας 31 όπου λέμε ότι είμαστε ότι είμαστε αντίθετοι με την μεταφορά ορισμένων δικαιωμάτων στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλληλείας που θα έχει αντικτύπωση σε ορισμένες τοπικές κοινότητες. Τώρα, αυτό το right-based management, δηλαδή διαχείριση βασισμένη σε δικαιώματα, είναι πολύ ανοιχτός ορισμός. Αυτός δεν είναι πολύ καλά ε, διευκρινισμένος. Μπορεί να σημαίνει ότι έχει κανείς μια άδεια αλίας και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η αλία και μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να ψαρεύει όσο θέλει. Δεν νοούμε δηλαδή αυτό. Θέλουμε λοιπόν εδώ να γίνει μια διευκρίνηση και έχουμε αλλάξει την παράγραφο 31 ώστε να λέει είναι αντίθετη με την υιοθέτηση από, ένωση, από την ένωση της μεταφοράς των ε, αδειών αλίευσης με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των τοπικών αλλιών κλπ. Αυτά είναι βασικά αυτά που συζητήσαμε. Ζητώ συγγνώμη και πάλι που δεν έχουμε νέες συμβαστικές τροπολογίες, αλλά όπως είπα, επ' αυτών εργαζόμαστε και θα τις υποβάλουμε όταν θα έχουμε την ευκαιρία. Και βεβαίω κάνουμε διάλογο και με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, αλλά θα συναντηθούμε και στην εβδομάδα του Στρασβούργου. Και μένω με ενδιαφέρον τώρα τι παρατηρήσει των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ, κύριε Λεβέν. Υπάρχει παρέμβαση από κάποιο συνάδελφο. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Επομένω, ε, να πω εγώ δύο λόγια, βάσει όσο είπε και η κυρία Λοβένα. Εμεί ε, αναμένουμε να υπάρχουν περισσότερε συμβαστικέ προτάσει που θα κατατεθούν. Είναι αλήθεια ότι σε μία πρώτη συνάντηση ε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες, όμως ορισμένοι συμβασμοί μένουν εκκρεμείς. Όχι μόνο για αυτό το πρώτο τμήμα, αλλά έχουμε και πολλού ε, άλλου συμβασμού που θα έπρεπε να κατατεθούν, να παρουσιάσουν στον επιτάπητο και νομίζω ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν κάποιε συμφωνίε ε, σε σχέση με την ποσότητα των τροπολογιών που παρουσιάστηκαν. Θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια λοιπόν και όπως είπε και η συγγήτρια να δούμε αν αυτή την εβδομάδα και αφού περάσαμε και ε, όλη αυτή την ε, τρελή κατάσταση με τις ψηφορίες σήμερα να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε περισσότερους συμβασμούς σε ένα έγγραφο που είναι λογικό. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Από ό,τι φαίνεται κινούμαστε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως. Ε, αν ε, τα είχαμε προγραμματίσει όλα μαζί, μάλλον θα μας έβγαινε. Έτσι, η συζήτηση, το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι με την κυρία Δαμανάκη. Δεν μπορούμε ε, να το κάνουμε νωρίτερα. Στις 5 θα συναντηθούμε με την κυρία Δαμανάκη και θα κάνουμε μια ένα μεγάλο διάλειμμα για καφέ και θα τα ξαναπούμε στις 5. Διακόπτουμε μέχρι τις 5 και θα συνεδριάσουμε για κλεισμένο των θυρών.